Ε, και κυρίως ε, για το χρονικό διάστημα μετά το 2015. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Έκλεισε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 8 ε, Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Προχωράμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γκόμες. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, έκλεισε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Συνεχίζει να είναι σβηστό το μικρόφωνο. Tratados. A política externa europeia deve η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ε, πολιτική εξωτερική η οποία ε, θα έχει συγκεκριμένες ε, πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερία. Θα πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτεί αυτή την πολιτική. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τις χώρες να πατάξουν τη διαφθορά και ειδικότερα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, δημόσιες ή ιδιωτικές, ε, γιατί αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Χρειάζεται να υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτού που κάνουμε εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξεκινήσουμε να αναρωτιόμαστε πώ είναι δυνατόν εμεί να Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε διαφθορά και ε, φυγή κεφαλαίων ε, πέραν, ε, σε τομείς πέραν της εκπαίδευσης. Θα πρέπει πραγματικά να σταματήσει το τραπεζικό απόρριτο το οποίο μειώνει τη διαφάνεια για την πραγματική διοκτησία των εταιριών, αποδυναμώνει την... θα πρέπει να ενισχύσουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως θα πρέπει επίσης να δώσουμε και δικαιοδοσία στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να αντιμετωπίσουν ζητήματα διαφθοράς ακόμα και αν λαμβάνουν χώρα εκτός ε, επικράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης ε, να ικανοποιήσουμε τους πολίτες οι οποίοι κατανοούν ε, πάρα πολύ καλά ότι η τρέχουσα κρίση και η αύξηση των χάσματος στην Ευρώπη μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων είναι αποτέλεσμα των ε, πολιτικών διαφθοράς ε, και της απορρίθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Η Ισπανία έχει πληγεί σοβαρά. Μετά είχαμε την ε, περίπτωση της ελληνικής υπόθεσης με τα υποβρύχια. Είχαμε γερμανικά υποβρύχια που αγοράστηκαν λόγω δωροδοκίας. Ε, αυτό ε, έγινε ε, και με εμπλοκή ανθρώπων από την Επιτροπή. Και τίποτα από αυτά δεν πήγε στα δικαστήρια. Πραγματικά βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητάνε από εμάς τους πολιτικούς να είμαστε ακέραιοι και να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε την διαφθορά στα κράτη-μέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Αυτό πρέπει να γίνει. Και δεν μπορούμε να πατάξουμε τη διαφθορά σε τρίτες χώρες αν δεν βάλουμε το δικό μας σπίτι σε τάξη. Θα πρέπει λοιπόν να προτείνουμε σειρά μέτρων. Πρώτα απ' όλα να εμπνευστούμε από τον νόμο Μπακνέξκι του Αμερικανικού Κογκρέσου που μιλάει για την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε έναν ε, μηχανισμό που να επιβάλλει κυρώσεις, ένα παρόμοιο μηχανισμό ε, για να υπάρχει πάγωμα των ε, παγίων στοιχείων οποιοδήποτε παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μην υπάρχει πρόβλημα με τους ακτιβιστές που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε τη διαφάνεια σε κάθε χώρα και ο κάθε οργανισμός που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και κάθε εταιρεία θα πρέπει να ονομάζει ποια είναι. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια δημοσιονομική, διότι ειδικότερα στις σχέση με τις τρίτες χώρες αυτό είναι απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα κατάλογο εταιριών που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην συμμετάσχουν σε διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον μέχρι να βάλουν το σπίτι τους σε τάξη. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο, έτσι ώστε οι χώρες, οι συγγνώμη, και οι χώρες να προωθούν την ακαιρεότητα. Τέλος, σε αυτή την έκθεση ζητούμε ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση όσων καταγγέλουν να ακούμε αυτούς που καταγγέλουν ότι χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκό χρήμα για τέτοιες διαφορεμένες πρακτικές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ε, θα φέρουν στο φως ε, τέτοιες περιπτώσεις ε, διαφθοράς. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκόμες. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία Catch και δίνω το λόγο στην κυρία Έλλη Τεστρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω να αρχίσω με ευχαριστίες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Είναι μια έκθεση που συνδέεται άμεσα με την επικαιρότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα, πρέπει να υιοθετήσει πιο απαιτητικού κανόνες. Και αυτό όχι μόνο στη δικιά της την επικράτεια, αλλά και να το λάβει αυτό υπόψη της και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες με τις οποίες έχει κάποια συνεργασία. Το έχουμε ήδη πει και το υπογραμμίζω ξανά ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οι ανισότητες, η κοινωνική αδικία είναι στοιχεία που βρίσκονται στη βάση της οικονομικής κρίσης με την οποία είμαστε σήμερα αντιμέτωποι. η απάτη, η διαφθορά, η απορρίθμιση του δημοσιονομικού τομέα μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε τώρα και αναγκαζόμαστε να κάνουμε τόσες θυσίες. Το γνωρίζουμε ότι οι πολίτες και η πολιτική τάξη έχουν πάρει διαζύγιο. Συνεπώς πρέπει να υιοθετήσουμε παραδειγματικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Είτε πρόκειται για τον δημοσιονομικό και οικονομικό τομέα, είτε πρόκειται για την πολιτική. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φερέιρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική, δεν μπορεί να αγνοεί την οτροπία που οδηγεί στις πρακτικές αυτές διαφθοράς. Τα διαφορετικά μέτρα που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα εφαρμόζουν στις χώρες της περιφέρειας, δηλαδή ιδιωτικοποίησης ή ιδιωτικοποίησης περιουσίας του δημοσίου, δημοσίων υπηρεσιών, το γεγονός ότι τελικά δεν υπερισχύει το κοινό συμφέρον, όλα αυτά οδηγούν στην ένδια. Και τελικά όλο και περισσότερες διασυνδέσεις υπάρχουν ανάμεσα στον οικονομικό και τον πολιτικό τομέα που οδηγούν σε διαφθορά και έτσι αποδυναμώνουν όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε για την πρόληψη. Και η πρόληψη περνάει από τη διακοπή τέτοιου είδους πολιτικών. Ευχαριστούμε. Κυρία Τόμα, συνεχίζω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως ε, Ευρωβουλευτής ε, από μια χώρα μετάβασης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και σε συνεργασία και ε, με άλλες χώρες, γιατί πρέπει να προστατευτούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι συνεργασία με χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση. Το αποτέλεσμα δεν θα εξαρτηθεί από την νομοθεσία, αλλά από τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, διαφθορά, αυτό πρέπει να το κάνει δικαιοσύνη. Σε χαμηλό επίπεδο διαφθορά είναι εξίσου σημαντική. γιατί με τον τρόπο αυτό διαχέεται σε ολόκληρο το σύστημα και έτσι καταλήγουμε σε εγκληματικέ πράξεις. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μήπως μπορεί να ανοίξει και το μικρόφωνο της Επίτροπος. Έχουμε λοιπόν ε, ζημιογόνες επιπτώσεις ε, στις κοινωνίες αυτό είναι κάτι που τον αγωνίζουν πλέον όλοι. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες ε, που ε, συνέταξε αυτή την έκταση. Η έκθεση της κυρίας Γκόμες πολύ σωστά επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει αξιόπιστη και να ασκεί ε, επιρροή στον αγώνα κατά της διαφθοράς εφόσον αντιμετωπίζει προβλήματα διαφθοράς, ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και οργανωμένου κλίματος στα δικά της τα σύνορα, στη δική της επικράτεια. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά αντιμετωπίστε ως ένα από τα πιο καθαρά τμήματα του κόσμου, αλλά και εδώ υπάρχει η διαφθορά. Επικύλει βέβαια και επεκτείνεται σε διάφορα κράτη-μέλη, εν πάση περιπτώσει αφορά όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τον Ιούνιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πακέτο κατά της διαφθοράς για την αντιμετώπιση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις των μελλοντικών δράσεων. Το πακέτο κατά της διαφθοράς ε, αναγκάζει την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της περισσότερο ε, σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ε, πολιτικής. Και θα ήθελα τώρα πιο συγκεκριμένα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που θίγει η έκθεση. Συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο να ρυθμίσουμε τις ε, δράσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για να γίνεται σεβαστός ο νόμος περί ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα είναι ο μόνος περιφερειακός οργανισμός που έχει εκφράσει την υποστήριξη του στο έγγραφο Monterey. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις ε, διαδικασίες ε, της διακυβερνητικής ομάδας των Ηνωμένων Εθνών ε, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός διεθνούς πλαισίου για το θέμα. Όσον αφορά την περίπτωση Μαγνίτσκι, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να έρθουν σε επαφή με αξιόπιστη ανάκριση, ανακριτή για να ε, διαλευκάνουν τα αίτια του θανάτου. Υπήρχαν κάποια στοιχεία που υποτίθεται έδειχναν, αποδείκναν γιατί πέθανε εκ των υστέρων και μετά θάνατον να καταδικάζεται η υπόθεση ο Μακνής αυτό είναι απαράδεκτο. Η Κομισιόν στράφει κατά του Μαγνίτσκι και του Λάουντερ μετά θάνατον ο κ. Μαγνίτσκι ε, χαρακτηρίστηκε ως εγκληματίας παρότι δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν έχουν διαλευκανθεί οι συνθήκες θανάτου του. Εμείς λάβαμε υπόψη μας τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που λένε να υπάρχει ε, μια πράξη, ευρωπαϊκή πράξη Μακνίτσκι. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι τα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Θα πρέπει οι κυρώσεις να χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο τελευταίας καταφυγής στο πλαίσιο μιας ε, ευρύτερης πολιτικής με διάλογο, συμπληρωματικές ενέργειες και άλλα μέσα. Αυτά απαιτούν το ύψιστο επίπεδο πολιτικής υποστήριξης και μπορούν να ε, προβλεφτούν μόνο εάν υπάρχει η ομόφωνη άποψη των ε, κρατών μελών. Κλείνει η συζήτηση. Αύριο την Τρίτη είναι η συζήτηση. Η ψηφορία με συγχωρείτε. Πάμε τώρα στην ε, έκθεση Ματσόνη.